Mes chers collègues, bonjour. Καθίστε συνάδελφοι, λέει η πρόεδρο. Να αρχίσουν. Avant d'ouvrir cette première Πριν αρχίσουμε αυτή μας την πρώτη συνάντηση της χρονιάς, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή χρονιά. γεμάτη εκπλήξεις, γεμάτη συναντήσεις, ανακαλύψεις, αλλά κυρίως υγεία και ευτυχία για σας και την οικογένειά σας. Ευχαριστούμε και καλή χρονιά και προς τους ε, διερμηνείς που τους έχουμε μαζί μας. Et Και επίσης να σας ευχαριστήσω όλους για το ότι είστε έτοιμοι για την τελική μας ευθεία φέτος. Αρχίζουμε τις εργασίες μας. Έχουμε τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτούς καλή χρονιά. Επίσης, καλώς όρισαν. Ε, και από ό,τι μου λένε, ο Βούλγαρος υπουργό είναι καθοδόν, είναι εδώ, όχι, όχι. Εδώ είναι, α. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ στην ε, Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Επομένω. πρώτον, έγκριση ημερήσια διάταξη. Το σχέδιο ημερήσια διάταξη, εγκρίνεται αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση. Δεν βλέπω να υπάρχει. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 15 η 21ης και 22 Νοεμβρίου του 2018 εγκρίνονται αν δεν υπάρχει ένσταση. Και για να ξεκινήσουμε με το δεξί, δεν έχω ανακοινώσει τη Πρόεδρου. Ευθύ αμέσω πάμε στο σημείο 4, το οποίο αφορά τον ε, μηχανισμό διασύνδεση τη Ευρώπη 14-20. Ε, την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και πρόκειται για τροποποίηση του κανονισμού 13-16 κάθετο 2013. Η συγκήτρια είναι υποφαινόμενη. Επομένως, On va pouvoir avoir un peu de silence. Merci. Ησυχία παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος. Όσον αφορά αυτή την έκθεση, πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω του σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ για τι τροπολογίε και ευχαριστώ για τη βοήθειά σα όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού που τροποποιεί αυτόν τον ε, διάδρομο Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος και από πλευράς ε, διασύνδεσης αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, Ιρλανδία σε περίπτωση που έχουμε σκληρό Brexit. Αυτό το σενάριο δεν είναι η αγαπημένη μας, η προτιμόμενη επιλογή ούτε της Επιτροπής μας, ούτε μου προσωπικά. Αλλά θα πρέπει να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, τους Ιρλανδούς πολίτες. Ε, γενικά το, το, των, θαλασσίων μεταφορών και τις ε, ακτές και επομένως η λογική είναι όταν υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά αυτές τις θαλάσσιες διαδρομές να προσαρμοστούμε. Επομένως Έχουμε τώρα τα, κάποια ζητήματα που είναι πρώτα πρώτα η συνέχιση της μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών σε σχέση με την Ιρλανδία και επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί σε μια ένωση των 27 ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και ε, ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο τέλος πάντων θα έχουμε καινούργια σύνορα και θα πρέπει να έχουμε ε, κάποιους λιμένες που θα γίνουν λιμένες για διεθνής μεταφοράς. Αυτά σε περίπτωση κάποιου Brexit χωρίς μεταβατική περίοδο. Σήμερα έχουμε το καλέ. 100% ασχολείται με τις ε, μεταφορές διαμέσου της μάχης, μάχης ως προς το και προς το Dover. Θα διαπιστώσετε στο κείμενο ε, ότι προσπαθούμε να διορθώσουμε διάφορα. Πρώτα μια ε, αντιστάθμιση όσον αφορά την, ε, την απώλεια σε κάποια λιμάνια γαλλικά λόγω των εξελίξεων και πρώτα πρώτα έχουμε το Δουνκέρκι, Λεάβρ, το Καλέ που εντάσσονται σε αυτό το διάδρομο Βόρειας Θάλασσας και οπότε θα αλλάξει αυτός ο διάδρομος και ο διάδρομος του Ατλαντικού και της Βόρειας και θα καλυφθούν οι, οι Βρέστη, το Σεν Λαζέρ, το Σερμπούρ, ε, Λεάβρ, Ρουέν και Παρίσι θα καλυφθούν από τη σχετική χρηματοδότηση και ήρθε η ώρα να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτά τα λιμάνια να αναπτυχθούν και επίσης να καλύψουμε και τις νέες ροές από την Ιρλανδία. Οπότε θα πρέπει να έχουμε σημεία τελωνιακού ελέγχου, ε, υγειονομικού ελέγχου, ε, κτηνιατρικού ελέγχου όσον αφορά τι συναλλαγέ με, με τον Βασίλειο που θα γίνει τρίτη χώρα. Και οπότε επιμένουμε στο θέμα του θα πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Αυτό να ισχύει πλήρως. Να μην αντιμετωπίζουν ε, τις συνέπειες της αλλαγής κατάστασης στα κράτη μόνα του. Και για αυτό και πρότεινα ε, εν είδη αντιστάθμισης για τα νέα λιμάνια για τους νέους ε, μεταφορείς και για όσους γενικώ θα φυγούν από το Brexit να υπάρξει κάποιο είδου ταμείο ε, κατεπήγων προσαρμογής εις το Brexit. Θέλω σε αυτό να με βοηθήσετε ούτως ώστε να προχωρήσουμε και να διαπραγματευτούμε τις ε, λεπτομέρειες, τα σχετικά ποσά με το Συμβούλιο. Αυτό για τους μεταφορείς μας, για τα λιμάνια μας, για τους διάφορους ε, φορείς να βρούμε για αυτούς ε, τους πόρους το ώστε να εξασφαλιστούν αυτού του είδους οι αντισταθμίσεις και έτσι οι σχετικές ροές να αντιμετωπιστούν γιατί θα μειωθούν αυτές οι ροές αν γίνει σκληρό Brexit. Οπότε πρόκειται για ένα σχέδιο κειμένου το οποίο διαπνέεται από τη λογική ε, το οποίο διαπνέεται επίσης από το ευρωπαϊκό πνεύμα όπως πάντα υποστηρίζω στην ε, ολομέλειά μας και ελπίζω να τα βρούμε και ελπίζω το κείμενο να ψηφιστεί, να υπερψηφιστεί με ευρεία πλειοψηφία. Και τώρα πρέπει να δώσουμε το λόγο στους ε, σκιώδεις εισηγητές. Κύριε Μιζελιέ, καλή χρονιά. Έχετε το λόγο. Το μικρόφωνο του ομιλητή σας ευχαριστώ για τόσα είπατε. Σας ευχαριστώ για το πνεύμα ε, που σας ε, διαπνέει και μας καλύψατε όλους ε, την ευγένειά σας και λοιπά. Στις 8 Ιανουαρίου είχαμε αυτή την συνάντηση πολύ παραγωγική ε, για αυτόν τον μηχανισμό, για την διασύνδεση σε περίπτωση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε 57 τροπολογίες, 6 συμβαστικές και πιστάει εκεί αντικαθρεφτίζονται οι θέσεις, ε, θέσεις της Επιτροπής και σήμερα έχουμε αυτό το σχέδιο κειμένο το οποίο καλύπτει σε αυτόν τον διάδρομο ε, Βόρειας Θάλασσας Μεσογείου τροποποιεί τον Ατλαντικό διάδρομο και καλύπτει τα γαλλικά ε, λιμάνια. Επομένως αυτό είναι καλά νέα και για τα λιμάνια και για την Ισλανδία. Ακόμα και σε την περίπτωση ενός σκληρού Brexit θα έχουμε κάποιες εγγυήσεις συνέχισης των ε, υπηρεσιών των σχετικών με τις μεταφοράς. Και, και εγώ ζητώ η Επιτροπή μας να υπερψηφίσει αυτές τις ε, τροπολογίες και έτσι ο κανονισμός να είναι έτοιμος, το σχέδιο του κειμένου έτοιμο το στις 29 Μαρτίου. Η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και η Καλή χρονιά σε όλους και όλους. Όπως ε, δηλώσατε ήδη, το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Συζητήθηκε σε μια επικοδομητική συνάντηση και για τον λόγο αυτό υποστηρίζω όλες τις συμβαστικές τροπολογίες που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία <coughs> σήμερα. Και παρακαλώ όλες και όλους να πράξουν το ίδιο, ώστε να έχουμε μια όσο γίνεται ευρύτερη πλειοψηφία, διότι βεβαίως είναι ζήτημα να διορθώσουμε κάτι που θεωρούμε ότι είναι ε, κάτι που ελισμόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ίδια κάναμε και στο πακέτο για, τους, για τις ε, οδικές συγκοινωνίες, οι μεταφορές. Και υπενθυμίζω τη θέση της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ ε, κυρία συνάδελφε. Κύριε Λόεν Γκριν, θέλετε να μιλήσετε τώρα. Εξ ονόματος της ομάδας σας ε, ECR. Ευχαριστώ πολύ και καλώς ήλθατε και καλή χρονιά. Η έκθεση εξ αρχής δεν ήταν αμφιλεγόμενη, συμφωνώντας με την ε, πρόταση της Κομισιόν. Μόνο τρεις τροπολογίες λάβαμε, για τις οποίες δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Ρονογκρίνη. Α, κύριε Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλή χρονιά σε όλους δεν θα παρατείνω με περιττό τρόπο την συζήτηση. Νομίζω ότι όλοι συμφωνήσαμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να υπάρξει απόλυτη δυνατή απόδοση ε, στις σχέσεις της ε, Ιρλανδίας με τους υπόλοιπους, αλλά να διορθωθεί και η κατάσταση των λιμένων. Μπορέσαμε να εξεύρουμε εύκολα ε, συμφωνία για τις έξι συμβαστικές τροπολογίες και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε όλες. Δεν θα υπάρξει εκ μέρου της ομάδας μας απολύτως κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ κύριε Ρικέ, λέει η πρόεδρος. Η κυρία Κλούνε. Ορίστε κυρία μου. Ευχαριστώ αγαπητή πρόεδρε. Καλημέρα και καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ για την δουλειά που κάνατε στον φάκελο αυτόν. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ορισμένα θέματα για τις ε, μεταφορές από Ιρλανδία προς ε, Υπηρετική Ευρώπη και υπάρχει πράγματι πολύ εμπόριο μεταξύ αυτών. Και βεβαίω η Ιρλανδία χρειάζεται να συνδεθεί και με τον Ατλαντικό διάδρομο, όπου δεν χρειάζεται, ε, δεν χρειάζεται έξτρα υποδομέ. Ε, χαίρομαι λοιπόν για το περιεχόμενο τη εκθέσεω. Έχω να πω και κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα σχετικό. Οι μικρομέσίε, ιδίω οι Ιρλανδικέ επιχειρήσει που χρησιμοποιούν τις ε, διαθαλάσσιε μεταφορές, για αυτές ο συντομότερος δρόμος είναι μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου. Εάν τελικώς αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, θα χρειαστεί να υπάρξει κάποια διασύνδεση μεταξύ Ιρλανδίας, ενό μέλους δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, της, και του λιμανιού του Καλέ, που είναι δηλαδή το κοντινότερο ε, υπηρετικό λιμάνι. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό να ληφθεί υπόψη στις σχετικές διαπραγματεύσεις για, το, για τις σχέσεις με το Ενωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ κυρία Κλούνε. Κυρία Μέισνερ, θέλατε να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Σύντομη παρατήρηση. Καλή χρονιά πρώτα. Η έκθεση είναι μια χαρά και συμφωνούμε με όλα. Αλλά επειδή είμαι και από φύση αισιόδοξη, η ευχή που θα κάνω για φέτος είναι να μην χρειαστεί η έκθεση και απευθύνω την ευχή αυτή σε όλους τους Βρετανούς που βρίσκονται στην αίθουσα. Ευχαριστώ κύριε Μέσνερ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα και εσείς κύριε Κόλσον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα, καλή χρονιά σε όλες και όλους του τους συναδέλφους σας. Χωρίς αμφιβολία δεχόμαστε ορισμένες τροπολογίες, 51 και 52, που επίσης και τις αντιστοιχούσες για τις αιτιολογικές σκέψεις που επιτρέπουν να περιληφθεί ένας αριθμός γαλλικών λιμανιών και ε, όπως ε, Καλέ, Δουνκέρκη αλλά και η Βερική Γάνδη στη ρύθμιση. Η πρόταση ξεπερνά την αρχική φιλοσοφία της πρότασης της Κομισιόν η οποία είχε την έννοια του κατεπήγοντος και όχι της προπαρασκευής και αλλάζει επομένως απολύτως την φιλοσοφία αυτού που ήθελε να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θέλω να πω για την έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζω ότι στην παρούσα εδώ ε, Επιτροπή είμαστε νομοθέτες. Ποιος είχε προβλέψει το Brexit στην πραγματικότητα κανείς. Άρα εγκύπτουμε στα νομικά θέματα. Και επειδή προσπαθείτε να με κάνετε να πιστέψω ότι το νομικό, η νομική πτυχή υπερισχύει της πολιτικής. Το ζήτημα είναι τι προσπαθούμε να διασώσουμε. Προσπαθούμε να διασώσουμε τις λιμενικές δραστηριότητες με τους φορείς που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα. Η θέση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να είναι όποια είναι, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να είναι διαφορετική. Και σας διαβεβαιώ ότι στη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου θα χρειαστεί να βρεθούν συμβιβασμοί μην προβάλλετε λοιπόν νομικά επιχειρήματα πριν να δείτε πρώτα-πρώτα την πολιτική διάσταση του θέματος. Σας ευχαριστώ λοιπόν, ωραία τα είπα. Ας συνεχίσουμε. Υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία της, ε, για την έκθεση μάλλον αυτή θα γίνει στις 10 το πρωί, 10 η ώρα. Συνεχίζουμε με το πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως, πρόταση για απόφαση ε, για την οδηγία 9653 σχετικά με προθεσμίες για ειδικούς κανόνες που έχουν σχέση με την ανώτατη διάρκεια αναπαύσεως στους θαλάμους οδηγήσεως ορισμένα θέματα αεροδυναμικής και ασφαλείας. Πάλι εγώ είμαι η συγκήτρια. Είναι η ημέρα μου σήμερα. Η οδηγία λοιπόν αυτή για τα μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα ε, θεσπίζει τις μέγιστες δυνατές ε, διαστάσεις για το εθνικό και διεθνές ε, για τη διεθνή κυκλοφορία. Η βελτίωση της αεροδυναμικής μορφής αλλά και των θαλάμων θα επιτρέψει να υπάρξουν σημαντικά κέρδη και για την ε, ενεργειακή απόδοση των ε, αυτοκινήτων, αλλά και για ε, την ασφάλεια στην κυκλοφορία. Πάντοτε για την 96-53 σχετικά με τις ανώτατες διαστάσεις των, των οχημάτων, είναι δυνατόν να γίνουν βελτιώσεις αυτές χωρίς να μειωθεί το ωφέλιμο βάρος των αυτοκινήτων. Η οδηγία προβλέπει ένα μορατόριο τριών ετών για την εισαγωγή αεροδυναμικών καμπινών θαλάμων διακυβέρνησης, δηλαδή θαλάμων οδήγησης και για τις σχετικές αλλαγές και τροποποίησεις σε ό,τι αφορά τις τεχνικές απαιτήσει για, την, για τις εγκρίσεις τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει προσαρμογή της οδηγίας ώστε να καταργηθεί το μορατόριο των τριών ετών και να μειωθούν οι προθεσμίες. Στο σχέδιο εκθεσιο μου εγώ προτείνω να προστεθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς τροποποίησης. Έως τώρα έχουμε λάβει τρεις τροπολογίες σχετικά με τον περιορισμό του συνολικού ανώτατου ωφέλιμου βάρους και για την ε, συνδρομική μεταφορά των οχημάτων αυτών και τις προθεσμίες. Θα συναντηθώ με τους και ηγητές τις επόμενες εβδομάδες και για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και η Επιτροπή Μεταφορών θα μπορέσει να ψηφίσει την απόφαση αυτή στις 22 πρώτου και να αρχίσει αμέσως τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Υπουργών τον Φεβρουάριο για το τελικό κείμενο υπό την επιφύλαξη ότι και το Συμβούλιο θα είναι διατεθειμένο να το πράξει. Να αρχίσουμε αμέσως την συζήτηση Πρώτα με τον κύριο Μαρινέσκου, ο οποίο είναι ο πρώτος και ο τη. Καλή σα μέρα κύριε Μαρινέσκου, καλημέρα κυρία Πρόεδρε. Πώς είστε. Θεωρώ ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι καλή. Να μειωθεί δηλαδή η προθεσμία για την εφαρμογή της οδηγίας. Νομίζω όμως ότι τέσσερις μήνες είναι υπερβολικά βραχία περίοδος. Οχτώ μήνες θα μας βοηθήσουν να αποφύγουμε οποιαδήποτε προβλήματα ανταγωνισμού μεταξύ εταιριών. Οχτώ μήνες νομίζω είναι η καλύτερη δυνατή περίοδος και έχω καταθέσει σχετική τροπολογία. Έχω και ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν μπορεί να δεχτεί την τροπολογία. Υπενθυμίστε τους ότι είναι επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, ότι έχουν καταθέσει πρόταση και ότι από τη στιγμή αυτή, που την καταθέτουν δηλαδή, νομοθέτες είναι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Δεν μπορούν να πούν ότι δεν μπορούν να δεχτούν την τροπολογία. Μπορεί να κάνουν μια πρόταση. Δεν μπορούν όμως να μην δεχτούν μια τροπολογία δική μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Είμαι βεβαία ότι έχει ακούσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί τις τροπολογίες. Η κυρία Ροβονταλόν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω μπροστά μου γραπτή την παρέμβαση του κυρίου Ασής που ε, κολλείεται. Ε, λέει ότι η ομάδα του σχετικά με τους κανόνες του μέγιστου μεγέθους του θαλάμου θεωρούν ότι θα επιτρέψουν να μειωθεί η κατανάλωση ενέργεια από τα φορτηγά αυτοκίνητα και θα βελτιώσουν την ασφάλεια. Δεν αναμένεται ωστόσο η επιτάχυνση τη ε, εφαρμογή να προκαλέσει προβλήματα για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Οι παρόντες κανόνε έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν την, ε, ε, το σχεδιασμό των νέων θαλάμων και δεν είναι υποχρεωτική. Για την πρώτη συζήτηση θεωρούμε ότι η μείωση του μορατόριου σε τέσσερι μήνε, όπω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι εύλογη και ε, λαμβάνει την υποστήριξή μα. Ευχαριστώ, κυρία Ροβονταλόν. Ο κύριο Λον Γκριν, θέλετε να λάβετε τον λόγο. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ήμουν λίγο αφηρημένο και δεν πρόσεξα καλά για το πρώτο θέμα. Ε, το σχόλιο μου λοιπόν αφορούσε το παρόν θέμα Ξέρετε ότι και ο ήλιος έχει κοιλίδες, άρα θα είναι εντάξει. Ξαναλέω πάντως και τώρα ότι η έκθεση δεν είναι αμφιλεγόμενη. Τρεις τροπολογίες δεν βρίσκω να είναι προβληματικές. Έχει καλός λοιπόν για μένα. Ευχαριστώ κύριε Λογκρίλ. Κυρία Μάισνερ, εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Συγγετρία. Συμφωνώ με τον Πέτερ Λόγκριν και λέγω κι εγώ ότι είναι ε, απολύτως μη αμφιλεγόμενη, μη αμφιλεγόμενη η έκθεση και επομένως μπορούμε να συμφωνήσουμε. Σεις κύριε Κράμερ τώρα, ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά και από μένα για όλες και όλους. Καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες. Πάντως για το παρόν θέμα, επειδή μιλήσατε και για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, το βάρος εκεί παίζει ένα ρόλο. Η γερμανική εμπειρία με τις διζελομηχανές πριν από 30 χρόνια ξεκίνησε επιδότηση για τις διζελομηχανές 18 λεπτά του ευρώ επιδότηση για κάθε λίτρο δίζελ. Διότι είχαμε πει τότε ότι οι μηχανές δίζελ καίνε λιγότερο και επομένως ε, είναι καλύτερο για το περιβάλλον. Όμως αυτό που κάνανε είναι να μεγαλώσουν τις μηχανές και τα αυτοκίνητα και επομένως αυτό το πλεονέκτημα ακυρώθηκε. Άρα το βάρος παίζει σημαντικό ρόλο. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω, ο κύριος Μαρινέσκο έχει βεβαίω δίκιο. Είμαστε κοινοβούλιο και ευρωπαϊκός νόμος εγκρίνεται μόνο εάν συμφωνήσουν και, οι τρεις, και τα τρία θεσμικά όργανα. Βεβαίω μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια σύντομη προθεσμία. Όμω και εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την, ε, το δικαίωμα να παρατείνουμε την προθεσμία. Εάν τώρα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι δεν το δέχομαι, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Είναι υποχρεωμένη να το συζητήσει όπω και εμεί συζητούμε την πρότασή τη. Ευχαρίστω να συζητήσουμε ισότιμα, όχι όμω κατ' εντολήν σα. Ευχαριστώ και καλή χρονιά και στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, πάντα. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Άλλος κανείς. Καλώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Ελίζαμπετ Βέρνερ. Καλή χρονιά και σε εσά Ελίζαμπετ. Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλες και όλους. Ευχαριστώ ιδιαίτερος εσάς κυρία Πρόεδρε ως εισηγήτρια του φακέλου, καθώς και τους και όλες εισηγητές. Λίγες τροπολογίες, πραγματικά πολύ λίγες, και αυτό μας ικανοποιεί, διότι φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει σημαντική συνένεση γύρω από τον φάκελο αυτό. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να διευκρινίσουμε προς τον κύριο Μαρινέσκου αυτό που είπαμε για την προθεσμία, για την θέση σε εφαρμογή ή μάλλον για την ε, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Νομίζω ότι υπήρξε κάποια παρανόηση. Ο στόχο μα είναι να γίνει αυτό το δυνατόν συντομότερο λόγω των ωφελημάτων που θα προσφέρει και στην αεροδυναμική μορφή των οχημάτων ε, καλύτερη ορατότητα, βελτιωμένη άνεση για τον οδηγό και θεωρούμε ότι αυτά τα ωφελήματα θα πρέπει να ε, γίνουν δυνατά το δυνατόν συντομότερο. Ε, τούτο λεχθέντος, ε, είμαστε απολύτως εύκαμπτες και εύκαμπτοι για να συζητήσουμε μια περίοδο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που να διευκολύνει. Δεν θα επιμείνουμε άκαμπτα στους τέσσερις μήνες. Είμαστε διατεθειμένες να συζητήσουμε κάτι, το, κάτι μακρύτερο, κάτι πιο ε, μια παράταση δηλαδή, της προθεσμίας αυτής, αρκεί να είναι λογική. Με την ευκαιρία θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα θέματα, τα οποία ίσως έχουν ε, σημασία σε σχέση με τις τροπολογίες κυρίας Αρνοτής. Ήδη σήμερα υπό την ισχύουσα νομοθεσία οι χώρες μέλη μπορούν να καθορίζουν για τις εθνικές μεταφορές το ανώτατο όριο. Οι 40 τόνοι αφορούν μόνο το διεθνές ή διαμεθοριακό εμπόριο. Και υπάρχουν βέβαια και ορισμένε χώρε μέλη οι οποίε έχουν υψηλότερα όρια βάρου για τι εθνικέ μεταφορέ. Οι εθνικέ αρχέ καλούνται να ελέγχουν ότι τα όρια βάρους γίνονται σεβαστά. Και οι αρμοδιότητες ελέγχου επίσης ενισχύονται. Υπάρχουν δύο αυτοματοποιημένα συστήματα μέσα στην οδηγία που προτείνεται και αυτά μπορούν, κάποια από τα δύο να επιλέξουν δηλαδή οι χώρε μέλη, θα γίνουν βεβαίω υποχρεωτικά πολύ σύντομα, ήδη το 2021. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι μάλλον ζήτημα εφαρμογής και ελέγχου και λιγότερο προσθήκης νέων διατάξεων. Τέλος, για τις διαδικασίες, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που μπορώ να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε και η Ρουμανική Προεδρία θεωρεί το ζήτημα αυτό ζήτημα προτεραιότητας και πρόκειται να ζητήσουν εντολή από τους μονίμους αντιπροσώπους για να αρχίσουν τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις πιθανώς αρχές Φεβρουαρίου και νομίζω ότι αυτό προσαρμόζεται καλά και με τον προγραμματισμό ψηφοριών σας στην Επιτροπή σας. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε ήδη από τον επόμενο μήνα να το προωθήσετε. Πρόκειται δηλαδή για ένα όριμο πλέον θέμα το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από τις ευρωεκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Βέρνερ. Όντω η ψηφοφορία επί τη εκθέσεω αυτή θα γίνει στι 22 Ιανουαρίου. Εκ παραλίλου ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο Υπουργών θα μπορέσει να καταλήξει σε θέση ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε τον τεμερή διάλογο αμέσω από τον Φεβρουάριο. Désormais, passons au point 6. Επομένως, τώρα ερχόμαστε στο θέμα υπαριθμών 6. Με εισηγήτρια την κυρία Κλούνε για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την δημιουργία ενιαίας θηρίδας για το θαλάσσιο εμπόδιο, θαλάσσιες μεταφορές για την οδηγία 2010-65. Ορίστε κυρία Κλούνε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ναι, καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω του σκιώδει για τη συνεργασία. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά εξαιρετική. Και μάλιστα από όλε τι πολιτικέ ομάδε, οι συμβιβαστικέ προτάσει θεωρώ ότι είναι ένα καλό μείγμα των θέσεων των ε, συνεισηγητών, των ε, σκιωδών εισηγητών και ξέρουμε λοιπόν πώς θέλουμε να προχωρήσουμε για το επόμενο ε, βήμα. 156 ήταν οι τροπολογίες που τέθηκαν, 10 οι συμβαστικές. Είναι καλή ισορροπία θεωρώ και πιστεύω ότι το θέμα αυτό της διευκρίνησης της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον και επίσης το γεγονό ότι προσπαθήσαμε να αυξήσουμε το επίπεδο της φιλοδοξία σε ό,τι αφορά το φόρτο που δέχονται οι πλεκτήτε, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει πολλή γραφειοκρατία ε, και πολλά συστήματα. Δεν θα τα αφαιρέσουμε, αλλά θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν πολλές αλλαγές για να εξασφαλίσουν ότι κάθε χώρα θα έχει μία ενιαία ναυτιλιακή αυτό υπήρχε σε κάποιες χώρες, αλλά τουλάχιστον να υπάρξει μια εναρμόνιση και στις υπόλοιπες ε, περιπτώσεις. Είναι τεχνικής φύσεως λοιπόν το ζήτημα αυτό. Δεν είναι πλάκι, είναι ιδιαίτερα η πολιτική χρειά. Και το θέμα είναι να βελτιώσουμε και την, ε, τα συνδικάτα, να βελτιώσουμε και να ενδρεμώσουμε το εμπόριο αυτό θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον όλων να υπάρξει η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση στον τομέα αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι θα υπάρξει υποστήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες και προσβλέπω στις περαιτέρω συζητήσει για το θέμα αυτό προκειμένου να το ολοκληρώσουμε εφόσον αυτό καταστεί δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λεκή Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την κυρία Κλούν και τώρα θα δώσουμε το λόγο Ο Φρέσκα Φεσκάστερ δεν είναι εδώ. Ούτε η κυρία Φώστερ. Η κυρία Μάιστνερ. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω την ε, κυρία Κλούν γιατί έχετε δίκιο. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή συνεργασία και θα συνεχίσει να είναι καλή η συνεργασία και στα πλαίσια του τρομερού διαλόγου και σε ό,τι αφορά αυτή την ενιαία ναυτιλιακή τρίδα, Όταν θα εφαρμοστεί, θεωρώ ότι θα διευκολύνει πάρα πολύ το ναυτιλιακό ε, εμπόριο και νομίζω ότι όλο ο κλάδο θα εγκρίνει την προσπάθεια αυτή. Ω εκ τούτου δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τι επερχόμενε διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ, κυρία Μάισνερ, λέει η Και τώρα το λόγο τον έχω εγώ, μια και είμαι και εγώ σκιώδης. Να σας ευχαριστώ, να σας ευχαριστήσω αγαπητοί συνάδελφοι για τη δουλειά που έκανε η κυρία Κλούν και ήταν καλή η δουλειά πραγματικά. Και δεδομένων και των συζητήσεών μας ε, στους ε, συντονιστές, στους ε, σκιώδησίτες, το κείμενο είναι τελικά καλό και πραγματικά έχει έρθει η στιγμή να δώσουμε μια πραγματική εναρμόνιση. Όταν μιλάμε για εναρμόνιση, εννοούμε για την εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασίων, για την εισαγωγή-εξαγωγή από ένα σκάφο, από ένα πλοίο σε χωρικά ύδατα της Ευρώπης. Επίσης, το θέμα των ε, μεταφορικών οδών και των αυτιλιακών οδών. Και έχετε δίκιο, κυρία Κλούν, στην Ευρώπη. Ένα φορτηγό που περνάει τα σύνορα χωρίς να αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, ενώ ένα πλοίο αντίστοιχα το οποίο φτάνει σε λιμένα αντιμετωπίζει ένα βαρύ γραφειοκρατικό άχθος. Και αυτό αποτελεί φόβητρο. Και πολλές φορές αυτό επαναλαμβάνεται και μέσα στους λιμένες του ίδιου κράτους. Αυτό λοιπόν καθιστά όλο τον ναυτιλιακό τομέα λιγότερο ανταγωνιστικό, πολύ λιγότερο ανταγωνιστικό από ό,τι άλλου. Και αυτό έχει επίση ε, αρνητικέ επιπτώσει και στις, ε, στον εργασιακό χώρο των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα αυτό και αντιμετωπίζουν όλε αυτέ τι ε, υποχρεωτικέ διαδικασίε. Θεωρώ λοιπόν την περίπτωση αυτή και είμαστε προ τη σωστή κατεύθυνση και θα βρούμε, θα καταφέρουμε να βρούμε έναν τρόπο για να ανταποκριθούμε και στα σημεία που είναι σημαντικά και στις προτεραιότητες και να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ κυρία Κλούν για τη δουλειά που κάνατε. Η κυρία Άντερσεν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δυστυχώ ο κύριο Κνούτ Φλέκενστάιν, ο σκιώδη τη ομάδα μου για την πρόταση αυτή, δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα. Έχει μια πολύ σημαντική συνάντηση στο Βερολίνο αλλά μου ζήτησε να τονίσω κάποια στοιχεία εξ ονόματο του. Καταρχά, να ευχαριστήσει την εισηγήτρια, την κυρία Κλούν και του υπόλοιπου κυρίε εισηγητέ για την πολύ καλή συνεργασία για το θέμα, για την πολύ ενεργή επικοδομητική συναντήση ε, μεταξύ των σκιωδών. Δεν υπήρχαν θέματα ουσιαστικά μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Έχουμε λοιπόν 10 καλού συμβιβασμού στην παρούσα φάση. Του υποστηρίζει οι σοσιαλιστέ και δημοκράτε και έχουμε καταθέσει και κάποιε τροπολογίε. Ω σκιώδη λοιπόν. Συγγνώμη κύρια Άντερσον, λέει η πρόεδρο Διακόπτη. Δεν είναι δυνατόν να παίρνετε το λόγο και να μιλάτε παράλληλα με μια συνάδελφο που μιλάει στο μικρόφωνο. Είτε θα δείξετε λοιπόν τον δέοντα σεβασμό και θα σιωπήσετε, είτε παρακαλώ να βγείτε από την αίθουσα. Και λυπάμαι κυρία Άντερσον που σας διακόψα έτσι απότομα. Άμα δεν είναι δυνατόν όμως να μην μπορούμε να σας ακούσουμε τελικά. Έχετε το λόγο και πάλι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος λοιπόν Φλέκενστάιν ε, εστιάστηκε σε τέσσερα βασικά στοιχεία στην έκθεση. Καταρχάς, εναρμόνιση μεταξύ διαφόρων μηχανισμών κοινοποίηση μεταξύ των κρατών μελών και λιμενικών αρχών, βασική προτεραιότητα του κανονισμού. Δεύτερον, ήδη φυστάμενα συστήματα τα, μάλλον τα ήδη φυστάμενα συστήματα επικοινωνία θα πρέπει να διατηρηθούν, γιατί έχουν γίνει σημαντικέ επενδύσει. Τρίτον, ε, εναρμόνιση με τα τελωνιακά συστήματα, λαμβάνοντα υπόψη και τι εξελίξει στο τελωνιακό τοπίο. Από, την, ε, από τις τυπικές διαδικασίες λοιπόν ε, των τελωνιακών συστημάτων δεν θα πρέπει να ξεκινήσει μια εναρμόνιση πρωτού λάβουμε υπόψη τι ήδη υφίσταται. Και τέλος, θα πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση όλου του εκπαιδευμένου προσωπικού για το θέμα τη ενία ε, θηρίδα. Είναι πολύ χρησιμοποιημένη η πρόταση. Την υποστηρίζουμε εμεί ω σοσιαλιστέ και δημοκράτε και η έκθεση θα αποτελέσει μια καλή βάση για του τρομερεί διαλόγου και μάλιστα με αρκετά ενωμένο τρόπο από πλευρά του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Άντερσον. Άλλο κανεί που θέλει να πάρει το λόγο. Κανεί. Άρα θα στραφώ προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσω το λόγο στην κυρία Κουσένσκα. Καλημέρα σας και καλή χρονιά σας εύχομαι. Καλημέρα Πρόεδρε, καλημέρα και σε εσάς κυρίε και κύριοι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους σας. Θα είμαι σύντομη. Καταχάσω. να ευχαριστήσω. Συγγνώμη, διακόπτη η πρόεδρο. Κύριε Μαρινέσκου, κύριε Αντελή. Αν θέλετε να τα πείτε, βγείτε έξω. Thank you. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε την εισηγητρία. Εξαιρετική δουλειά καθ' όλη τη διαδικασία και του κοιότης ασφαλώς. Και όλη την Επιτροπή να ευχαριστήσουμε για την κατανοή και τη χρονική πίεση υπό την οποία βρισκόμαστε. Ξέρω ότι έχετε ε, διεκπαιρεώσει αυτή την έκθεση σε χρόνο ρεκόρ για να μπορέσουμε να πετύχουμε στα πλαίσια του τρομερούς διαλόγου μια συμφωνία ε, είναι μια σαφής ένδειξη του ότι κατανοούμε εξαιρετικά των βασικών, της βασικής προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να διευκολυνθεί η μεταφορά προϊόντων, το θέμα της εναρμόνισης, σε ό,τι αφορά τη κοινοποίηση των τοπικών αυτών διαδικασιών. Ήταν στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας όταν υποβάλαμε την πρόταση αυτή. ορίζω λοιπόν την αναγνώριση του θέματος αυτό στην έκθεση και ιδιαίτερως στις 10 συμβιβαστικές τροπολογίες που κατατέθηκαν μετά από τη συνάντηση των σκιωδών. Να καλωσορίσω επίσης την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενισχυθεί η αρχή μιας ενιαίας ε, ομάδας ε, πληροφοριών και ενός ενιαίου μηχανισμού για να μην υπάρχουν ε, περιττές ε, διαδικασίες και προδιαγραφές ε, για την ε, διάδοση των πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό λοιπόν σχετίζεται με την αποτελεσματική και αποδοτική εναρμόνιση των τυπικών αυτών διαδικασιών. Επίσης υπάρχει και πρόταση του Κοινοβουλίου για την αμφίδρομη επικοινωνία που θα διευκολύνει τη διαδικασία και θα μειώσει το γραφειοκρατικό άχθος και την όλη διαδικασία γενικότερα. Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία επιβάλλει το Κοινοβούλιο τα οποία θεωρώ ότι θα τα διευκρινίσουμε στον τριμερή διάλογο, είμαι σίγουρη, προκειμένου και ο πολιτικό στόχο του Κοινοβουλίου να εκπληρωθεί και να βελτιώσουμε ενδεχομένω κάπω ε, την διατύπωση. Ένα λεπτάκι επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε αυτά. Ε, Καταρχά, σε ό,τι αφορά την τεχνολογική ουδετερότητα, μια πολύ σημαντική αρχή που υπογραμμίζει οτιδήποτε έχει να κάνει με την καινοτομία και τι καινοτομικέ ε, τεχνολογίες. Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την εναρμόνιση και για την ψηφιακή αναφορά και την εναρμόνιση που θα αποτρέψει και πάλι ανάπτυξη διαφορετικών συστημάτων με διαφορετικές τεχνολογίες. Αυτό αντίθετα θα στραφεί, θα αποβεί προς την εναρμόνιση. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο αναφέρθηκε από την κυρία Άντερσον, το θέμα των υφιστάμενων διόδων επικοινωνία λαμβάνουμε ασφαλώς υπόψη πλήρως το γεγονός ότι τέτοιες, τέτοια κανάλια επικοινωνίας είχαν ήδη δημιουργήσει από εθνικές αρχές, από τους λιμένες, αλλά παράλληλα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιείται μία οδός επικοινωνία για την αναφορά στοιχείων. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε με το ενιαίο τέτοιο περιβάλλον και την ενιαία θηρίδα. Καταλαβαίνω λοιπόν ε, την ε, πολιτική επιχειρηματολογία που κρύβεται από πίσω από την πρόταση αυτή. Ελπίζω στα πλαίσια του τριμερού διαλόγου να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε μάλλον να βρούμε έναν τρόπο που δεν θα μας οδηγήσει τελικά στη συνύπαρξη πολλών διαφορετικών συστημάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ λοιπόν και πάλι κυρία Κλούμ να ευχαριστήσω για τους Χιώδης. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας στα πλαίσια του τριμερού διαλόγου. Ευχαριστώ, λέει και Πρόεδρο. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι απαντήσει που μα έδωσε και να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κλούν για να συνοψίσει. Μάλιστα, να πω δύο λόγια. Να ευχαριστήσω όλου όσοι πήραν το λόγο. Πολύ θετικά τα όσα ακούσαμε σήμερα το πρωί. Να μην σα ζωρίσω παραπάνω, να πω σε ό,τι αφορά αυτά που μόλις μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι. Καταλαβαίνω ότι εννοείται ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την διατύπωση. Το θέμα είναι να αποτυπώνεται και η φιλοδοξία, το επίπεδο φιλοδοξία των βουλευτών και του Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικό φυσικά να υπάρχει μια κάποια εναρμόνιση. Θα πρέπει να έχουμε ε, μια βασική εναρμόνιση. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέπει την τεχνολογία. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε στον τρεμερή διάλογο μια σωστή ισορροπία και ελπίζω να καταλήξουμε τάχιστα στο σημείο αυτό της Εξέβρεση της συμβαστικής έτσι, αυτή λύσης. Από πλευρά μα σκοπεύουμε να προχωρήσουμε το φάκελο αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για να καταλήξουμε στη θέση μα για το τριμερή διάλογο. Έχουμε πλέον δασμεύσει από όλε τι πλευρέ. Ελπίζω να καταφέρουμε πριν από το τέλη τη θητεία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και του Κιόντι και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλη την υποστήριξη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λαϊκή Πρόεδρος. Να υπενθυμίσω ότι η έκθεση αυτή θα ψηφιστεί σήμερα. Μάλιστα, Πρόεδρε. Έχουμε λοιπόν ε, έχουμε προχωρήσει πολύ γρήγορα και γι' αυτό λοιπόν να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 10 λεπτών.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναλέει ο πρόεδρος. Παρακαλώ κύριε Μαρινέσκου. Η κυρία Φώστερ. Κάποιος, συνάδελφοι, ξέχασε ένα ποντίκι, ένα ποντίκι Χιούλετ Πάκαρντ εδώ στο έδρανό μου. Ε, όπου βιασύνη έφυγε ξεχνώντας το... Οπότε εδώ είναι αν θέλει να το μαζέψει. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε εμείς κύριε Φώστερ λέει ε, οπότε να έχουν, έχει απολεστεί αυτό το ποντίκι υπολογιστή. Και τώρα ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας. Πριν αρχίσουμε τις ψηφοφορίες μας, καλωσόρισαν όλοι αυτοί οι συνδικαλιστές. Ένα σωρό σήμερα. Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Θα κάνουμε ένα τεστ, μια εικονική ψηφοφορία για να δούμε αν έχουμε απαρτία κλπ. Ψηφίζουμε. Ένας παραπάνω ψήφισε για το ΕΛΚ. de trop. Deux, Δύο, δύο παραπάνω. Διορθώνει η γραμματεία. Δύο παραπάνω για το ΕΛΚ. Ας κάνουμε άλλη μια δοκιμή, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε. Πολύ ωραία. Διορθώθηκε. Μπράβο στο ΕΛΚ. Προς το παρόν, καλά τα πήγατε. Α, τώρα όμως ξαναψήφισε ένας παραπάνω. Il ne doit pas voter. Il y en Ένα παραπάνω ξαναλέει πρόεδρο για το ΕΛΚ. On ne peut pas commencer s'il y a un en plus. On attend. Maintenant c'est OK. Maintenant c'est OK. Τώρα εντάξει, λέει ο γραμματέα. C'est bon pour le... Εντάξει, το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο εσείς. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Ζλωτόφσκι. Θέλω να σας ενημερώσω για το εξής. Στις μεταφορές έχουμε κάποια εκδήλωση διαμαρτυρίας από Εστονία, από τις τρεις από τις βαλτικές χώρες και από Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία και θα ήθελα αυτό να σας γνωστοποιήσω ότι έχουμε αυτή την εκδήλωση διαμαρτυρία. τώρα, την ώρα που εμείς εδώ συζητούμε. Η διαμαρτυρία αφορά ε, ένα θέμα από αυτά που θα ψηφίσουμε και θεωρείται ότι Εάν περάσει το θέμα το οποίο ψηφίζουμε, θα οριστικοποιηθεί το χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Δεν θα υλοποιηθεί η κοινή αγορά για την οποία φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, λέει ο Πρόεδρος. Να σας πω το εξής. Αυτό το πακέτο για την κινητικότητα έχει κάνει μια διαδρομή πάνω από ένα χρόνο και σήμερα ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας. Εμεί μου λέτε ότι θα πρέπει να αναβάλουμε την ε, ψηφοφορία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένταση από πλευρά των εργαζομένων. Αλλά εμείς είμαστε νομοθέτες και ρόλος μας είναι να βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας τους. Ήρθε τώρα η ώρα να ψηφίσουμε και έκαστος εξημών αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν μπορείτε να με εκβιάσετε ότι χρειαζόμαστε χρόνο, δεν είμαστε έτοιμοι. Ε, όχι. Ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας. Allez. Monsieur Marinescu. Έχει το λόγο ο κύριος Μαρινέσκου. Ένα λεπτό έχετε κύριε Μαρινέσκου. Ευχαριστώ πολύ. Χθες βράδυ Σα διαβιβάσαμε έτοιμα αναβολή τη ψηφοφορίας γιατί δεν υπάρχει μετάφραση, διερμηνία τέλος πάντων προς όλες τις ε, γλώσσες όπου αφορούν κάποιες εναλλακτικέ ε, ε, συμβαστικέ τροπολογίες. Νομίζω ότι είναι σαφής η διάταξη που λέει ότι πρέπει να λειτουργεί η ψηφοφορία. Δεν μπορείτε να πείτε όχι. Μπράβο στην γραμματεία που δούλεψε μέρα και νύχτα, αλλά δεν ολοκληρώσανε. Άρα έχουν πρόβλημα με, με, με τα κείμενα. Τα κείμενα, τα μετάφραση, όχι δερμηνή, μετάφραση. Δεν έχουμε όλα τα κείμενα, επομένω δεν μπορείτε να μα πείτε όχι, γιατί αυτό είναι διάταξη του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Και έχετε αντιστρέψει ε, τα θέματα, έχετε αντιστρέψει τη σειρά της ψηφοφορίας και πρώτα θα πρέπει ε, να μας πείτε ότι θέλατε να ψηφίσουν πρώτα των ε, εισηγητών της συμβαστικές, αλλά θα πρέπει να εφαρμόσετε διάταξη και να αναβάλλετε. Κύριε Μαρινέσκου, όχι δεν δέχομαι αυτό το οποίο είπατε, ε, το ότι δεν σέβομαι τον κανονισμό. μέσα στη νύχτα όλα μεταφράστηκαν σε βουλγαρικά, ουγγρικά, πολωνικά κλπ. Έγινε μετάφραση. Ένα αυτό. Δεύτερον, κάτι άλλο το οποίο είναι απαράδεκτο και σας το τονίζω ότι εσείς ήσασταν εισηγητή για την αεροπλοεία. Τι έγινε με τι μεταφράσεις εκεί. Ε, δεν είχαν μεταφράσει τα κείμενα στι αντίστοιχε γλώσσε και κάναμε τη δουλειά μα με τα αγγλικά. Και τώρα τι μου λέτε, κάνατε ένσταση ότι δεν είχατε έγκαιρα την μετάφραση και ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Ε, όχι, αυτό που λέτε δεν στέκει. Υπάρχουν και όρια. Σας το τονίζω. Να αναλάβει έκαστος τις ευθύνες του θα ψηφίσουμε. Δεν θα συνεχιστεί η συζήτηση. Κυρία Κυραπίνη, θέλετε το λόγο. Έχετε μισό λεπτό. Τριάντα δευτερόλεπτα. Επανειλημμένα έχουμε ενστάσεις βάσει του κρονισμού για έλλειψη μετάφρασης. Και το έχει γίνει αυτό και για μία μόνη γλώσσα, τα πορτογαλικά. Επίσης δεν μπορεί να μας πείτε ε, Τότε με ότι υπάρχει αυτή η προθεσμία ενώ δεν υπήρχαν ακόμα οι μεταφράσεις και αν τις κάνετε το, το, το, τα μεσάνυχτα αυτέ τι μεταφράσει. Το ανάποδο θα πρέπει να γίνεται. Πρώτα να έχουμε τις ε, μεταφράσει και ε, να πάμε στις ε, συμβαστικέ βάσει του μεταφρασμένου κειμένου. Ανα, αντιστρέψατε την σειρά των πραγμάτων. Δεν είναι στο, είναι ντροπή. Πρόεδρος. Εγώ δεν συνεχίζω σε αυτό το πνεύμα. Ολοκληρώσαμε. Δεν είναι το θέμα μας τώρα. Η μετάφραση αυτό γίνεται πολλές φορές και στην Ολομέλεια. Να έρχεται η μετάφραση μία ώρα πριν τη συζήτηση. Ξέρω τη διαδικασία. Μην με κατηγορείτε. Ψηφίζουμε τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Μαρινέσκο. Συγγνώμη, πρόεδρε, αλλά θα πρέπει να σεβαστείτε τον κανονισμό. Αυτό το παράδειγμα που είπατε για τον ε, κείμενο που εγώ είχα εισηγηθεί της ΙΑΣΑ δεν ε, προσφέρεται. Γιατί τότε για την ΙΑΣΑ κανείς δεν είχε ε, προβάλει ένσταση. Τώρα προβάλλουμε ένσταση επικαλούνται τους κανόνες. Ναι, ναι, ναι, ναι, τηρούνται οι κανόνες. Αν δεν θέλετε να συμμετάσχετε στην ε, ψηφοφορία, ε, αναλάβετε την ευθύνη σα. Και δεν θα λάβει άλλο το λόγο. Ψηφίζουμε αμέσως τώρα. Πρώτον, πάμε στην ψηφοφορία και δεύτερον, δεν δέχομαι το επιχείρημά σας, γιατί έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος που μας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα. Και τι μου λέτε την τελευταία στιγμή δεν έχουμε μετάφραση. Αρκετά. Πάμε στην πρώτη έκθεση. Έκθεση κιλώνεν. Αφορά την απόσπαση εργαζομένων. Αρχίζουμε. Nous passons tout d'abord au compromis. Πρώτα, Πάμε στη συμβαστική της εισηγήτριας. Κι Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για επαλήθευση. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. C'est bon, c'est correct. Καλώς. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Nous ne sommes pas là au Κοιτάξτε, δεν είμαστε εδώ για να δίνουμε θέαμα. Δείξτε λίγη υπευθυνότητα. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Εναλλακτική, συμβαστική, ε, υπέρ. Κύριε Κουρουμπάτσεφ, έχετε μισό λεπτό. Έχω μία πρόταση, κ. Κουρουμπάτσεφ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Να μην το κάνουμε, μην κάνουμε την ψηφοφορία με ανάταση της χειρός, αλλά ηλεκτρονικά. Νομίζω και για τα τρία αυτά θέματα, μια που είναι σημαντικά. Όλα ε, ηλεκτρονικά. Νομίζω και εσάς ωφελεί η Πρόεδρε και έτσι υπάρχει και ευξημένο κύριο στην ψηφορία η Πρόεδρος. Δεν έχω πρόβλημα. Ας τα ψηφίσουμε όλα, όλες τις εναλλακτικέ συμβαστικές ε, ηλεκτρονικά. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, να το κάνουμε έτσι. Συνεχίζουμε. Η εναλλακτική ε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική, εναλλακτική, α. Ψηφίζουμε. Je ferme le vote. Πέρα τη εφορία. Εναλλακτική συμβαστική σε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτονται. Εναλλακτική συμβαστική B. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτονται. Ντε. Εναλλακτική συμβαστική Ντε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. F. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Il est convenu. Περαδόθηκε η ψηφορία. Τελίνσκα, μισό λεπτό. Δεν θέλω να ανοίξω τη συζήτηση, κυρία Πρόεδρε, λέει ο Τέλινσκα, αλλά βλέπουμε τώρα ότι ένα από τα τρία μέρη του πακέτου δεν τα κατάφερε να περάσει την ψηφοφορία. Θα σας παρακαλέσω να μας δώσετε 10 λεπτά διάλειμμα για συνεννόηση, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το γεγονός έχει απήχηση στις άλλες δύο προτάσεις. Θα χρειαστεί λοιπόν να γίνει διαβούλευση εντός των πολιτικών ομάδων, αλλά θα σας παρακαλέσω επίσης να επιτρέψετε να γίνει μια σύντομη συνάντηση Προέδρου και Συντονιστών. Η Πρόεδρος, κύριε Τελίτσκα. όταν μια έκθεση του πακέτου των, της κινητικότητας, όπως συμβαίνει τώρα, δεν εγκρίνεται, πρέπει να συνεχίσουμε την ψηφοφορία για να δούμε τι θα κάνουμε στην συνάντηση των συντονιστών για το σύνολο των εκθέσεων. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την έκθεση. Όπως είπα ήδη, το πακέτο της κινητικότητας είναι πακέτο το οποίο ε, θα γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τρεις πτυχές. Αρκεί να ιτηθεί στην ψηφοφορία η μία, ώστε να μην μπορούν να συζητηθούν οι άλλες δύο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και επειδή βρισκόμαστε στην συζήτηση θα δώσω πολύ σύντομα, 30 δευτερόλεπτα, τον λόγο στους συντονιστές. Ο κύριος Βιμ Βαντεκάμπ. Κυρία Πρόεδρε, δέχομαι την πρότασή σας. Νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία. Όλο το κοινό σε όλες τις χώρες στην Ένωση οι εργοδότες θέλουν να γνωρίζουν τι θα γίνει. Αν αναβάλουμε τώρα, η εικόνα είναι εντελώς ασαφής και θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ο κύριος Ερτούγκ. Το ίδιο. Συμφωνείτε λοιπόν. Η κυρία Κιλένεν. Το ίδιο. Κύριε Κράμερ. Εγώ ήθελα να πω ότι γνωρίζουμε ότι είναι περίπλοκη η διαδικασία. Στο σύνολό της. Τα έχουμε συζητήσει. Έχουμε θέση. Τώρα καλούμεθα να ψηφίσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν, λέει η Πρόεδρος. με την έκθεση Van de για τις συνθήκες εργασίας, κοινωνικές συνθήκες, ελάχιστο όριο ε, ανάπαυσης και χρόνων ανάπαυσης. Είστε έτοιμοι? Η συμβαστική του εισηγητού. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συνεχίζουμε. Συμβαστική Β. Εναλλακτική. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Αυτό θα γίνει τώρα με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική δέλτα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την συμβαστική δέλτα, D. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική σε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική α. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη και αυτή. Συμβαστική ε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη ομοίως. Δηλαδή η έκθεση του κυρίου Βάντε Κάμπ, όπως και της κυρίας Κιλένεν, δεν εγκρίνονται. Προχωρούμε στην έκθεση του κυρίου Ερτούκ. Σας παρακαλώ. Συμβαστική του εισηγητού. Ψηφίζομαι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η συμβαστική του κύριου Ερτούγκ εγκρίνεται. αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Προσκαλώ τους συντονιστές μετά την ψηφοφορία σε συνάντηση για να συζητήσουμε τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε. Για τις συνέχειες, μάλλον για τη συνέχεια και τις επιπτώσεις του πακέτου κινητικότητας. Και συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Έκριση Del Σας παρακαλώ λίγη ησυχία ακόμα, δεν έχουμε ολοκληρώσει τις ψηφοφορίες. Αν επιθυμείτε να... Κυρία Παρπαντέλ, τηλέφωνο έξω. Κυρία Ντελμόντε, ψήφι υπέρ, άρθρο 1, παράγραφος 1. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Ψηφίζουμε τελική ψηφοφορία της εκθέσεως αυτής. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Η έκθεση κυρίας Ντεμόντε εγκρίνεται. Διαπραγματευτική εντολή. Ψηφοφορία για τη διαπραγματευτική εντολή. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Κυρία Ντεμόντε, προετοιμαστείτε διότι θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Και μπράβο σας. Συνεχίζουμε. Ε, με την έκθεση της κυρίας Ντελή. Τροπολογία 6. Υπέ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία παριθμών 9. Αρχίζει η ψηφοφορία. Σας παρακαλώ ισχύα. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές αποτέλεσμα ασαφές γι' αυτό θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει τροπολογία 56 πέρας Μου φαίνεται ότι ήσασταν κουρασμένοι και δεν σηκώσετε τα χέρια. Εγκρίνεται πάντως. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνούμε αμέσως στην τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέζι 1 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προχωρούμε αμέσως στην τροπολογία 2 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρινεται Ένα 1α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ συμβαστική 2 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέζι πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτή τη φορά. Πέρας. Ψήφι υπέρ 45. Ούτε μία κατά. Δύο αποχές. Η έκθεση της κυρίας Ντελή εγκρίνεται για την διαπραγματευτική εντολή με Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τμήμα αυτό των θαλάσσιων μεταφορών του Brexit. Αρχίζει η ψηφοφορία για τη διαπραγματευτική εντολή. Πέρας. Εγκρίνεται με ουδεμία ψηφοκατά και ουδεμία αποχή. Συγχαρητήρια, κύριε Ντελή. Ας συνεχίσουμε. με την έκθεση Κλούνε. Ας αρχίσουμε. Τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική δηλαδή. Τροπολογία 60. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Κύριε Υπουργέ, θα τα ξαναπούμε στην Επιτροπή μας. Α, αποχαιρετά τον Βούλγαρο Υπουργό. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Θέλετε επαλήθευση. 67. Ωραία. Αρχίζει ηλεκτρονική επαλήθευση για την 67. Αρχίζει. Πέρας. Απερίφθη. Είχατε δίκιο κύριε Βαντεκάμπ. Βέβαια δεν έχετε πάντα δίκιο. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 3. Εγκρίνεται. Προχωρούμε αμέσως στην συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες, 143 και 29. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Δύο ταυτόσημες τροπολογίες, 142 και 29. Εγκρίνονται και με μεγάλη πλειοψηφία. Συνεχίζουμε. Τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες. 144 έως 146. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Δύο ταυτόσιμες. 147 και 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 149. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 150. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κύριε Βαντεκάμ, δεν ψηφίσετε καν τις δικές σας τροπολογίες. 153. <clears throat> Υπέρ. Α, μάλιστα, τώρα ναι. Κατά αποχές. Δεν είναι σαφές όμως το αποτέλεσμα. Θέτω σε ηλεκτρονική ψηφοφορία την 153. Νομίζω όμως ότι εγκρίνεται. Για να δούμε. Πέρασε. Σαφέστατο το αποτέλεσμα, είχατε δίκιο. Συνεχίζουμε. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 30 υπέρ. Κατά αποχές Δεν είπα καν ακόμη αν εγκρίνεται ή όχι και μου λέτε ήδη ότι θέλετε επαλήθευση. Καλά. Ας επαληθεύσουμε. Τροπολογία 30. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά Αποχέ. απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά Αποχέ. δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 51 εκπίπτει, η 50 ομοίως, της κυρίας Ντελή επίσης εκπίπτει. Δύο ταυτόσημες τώρα, 53 και 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, στο σύνολό της η έκθεση, η ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει, πέρας, με μεγάλη πλειοψηφία έγκριση. Συγχαρητήρια κυρία Κλούνε. Και ψηφίζουμε αμέσω και την διαπραγματευτική εντολή ώστε να μπορεί να αρχίσει η διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Αρχίζει τις προετοιμασίε, κύριε Πλούνε, αρχίζει η διαπραγμάτευση. Σας ευχαριστώ. Και να περάσουμε λοιπόν τώρα στην έκθεση του ενός και μοναδικού Ντομινίκ Ρικέ. Για τα μέτρα εξορθολογισμού για τα δίκτυα TNT. Καλά τα λέει Ντομινίκ. Τέλεια. Να ξεκινήσουμε. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Έγκρινεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Έγκρινεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Έγκρινεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Εντάξει, το βρήκατε το συμβαστικό Κείμενο τη 7. 7 λοιπόν, η συμβαστική υπέρ. Κατά. Απόχε. Έγκρινεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Απόχε. Έγκρινεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. απόχε. Έγκρινεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Απόχε. Έγκρινεται. Στι συντολογικές σκέψει. Πάμε τώρα. Τη Επιτροπή. 36 μάλλον. Τροπολογική 36. Υπέρ. Κατά. Απόχε. Απορρίπτεται. Ρέτζ 15. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. Και τώρα να ψηφίσουμε το σύνολο της έκθεσης. Ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. 35, 37 υπέρ. 6, 6 κατά. Συγχαρητήρια στον κύριο Ρικέ. Εγκρίθηκε η έκθεσή σας. Και συνεχίζουμε με την έκθεση Allez, nous commençons. Qui concerne, bien sûr. Κύριε Φαμίτελμπριχ, για τις προτάσεις, για τις σχετικέ διτάξει έγκριση τύπου για μηχανοκίνητα οχήματα σε ό,τι αφορά τη γενική του ασφάλεια. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Unblock. Ε, ψηφίζουμε την 4275 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 43 και η 80 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άλλε δύο, 48 και 49 υπέρ. Ταυτόσιμε. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνονται. Να κάνουμε μια επαλήθευση για τι δύο αυτέ τροπολογίε, 48 και 49. Παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Η 51 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 50. Α, καταπληκτή. Συμβαστική 10 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. Υπάρχουν ενστάσεις κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Θα την ψηφίσουμε. Unblock. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας κάνουμε μια επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε, λέει η Πρόεδρο, την προφορική τροπολογία. Την 58 και την 88 από κοινού. Γι' αυτό και είναι on block. Πέρας ψηφοφορίας, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 65. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Έλεγχος. Κύριε Φώστερ. Ναι, ένα σύντομο σημείο να δείξω. Αντί να λέμε τσεκ από πλευρά των ομάδων ή ατομικά, να ζητήσω από τους συντενιστές να μας ε, υποδεικνύουν ε, τι γίνεται σε κάθε ομάδα, για να μην χρειάζεται να ζητάμε κατά τέτοιο λίγο έλεγχο. Και για σας φαντάζομαι ότι είναι λίγο πιο εύκολο. Ναι, ναι, αλλά βέβαια σηκώσετε καλά το χέρι σα, ε, Βίμ. Πού να ξέρω κι εγώ. Κυρία Φώστερ, λέει η πρόεδρο. Ο κύριο Βίμ μου προφανώ και δεν σηκώνει καλά το χέρι του. Το είπα κι εγώ προηγουμένω. Αλλά ενδεχομένω ε, αυτά που λέει ο συντονιστή να μην τα ακολουθεί ο καθένα μέσα στην πολιτική ομάδα και σε αυτό θα χρειαστεί να προσέξουμε. 66 παρακαλώ, υπέρ. Έλεγχος ζητήθηκε. Συντήθηκε έλεγχος για την 65 παρακαλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Έναρξη. Για την 65. Πέρας. Εγκρίθηκε. Α, σας το έλεγα, δεν πιστεύατε. Συνεχίζουμε. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Καταπίπτει, συγγνώμη. 68. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Νομίζω ότι Εγκρίνεται, αλλά κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 68, παρακαλώ. Έναρξε. Και πέρας τώρα. Απορρίφθηκε. Unblock 69, 177, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφέ. Η 70 παρακαλώ. Ψηφίζουμε την 70. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Θέλετε να επαληθεύσουμε την 89. Ε, Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Για μένα το αποτέλεσμα είναι σαφές, αλλά εν περιπτώσει. Αφού το ζητάτε. Πέρας. Γιατί κάνουμε την επαληθεύση, γιατί το δικαιούστε. Δεν μπορούμε να είμαστε αντιδημοκρατικοί, κύριε Βίμ Κάμπ. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 2. Υπέρ. Α, συγγνώμη. Η Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και περνάμε στη συμβαστική περιθμόν 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 134. Unblock. 135, 169, 170. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Πέρας. Απορρίφθηκε. Δύο ταυτόσιμες τροπολογίες, η 151 και η 152, υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. Ε, unblock τώρα, 153, 154, 173, υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίφθηκε. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Δύο ταυτόσιμες. 158 και 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, παρακαλώ. Ηλεκτρονικά να κάνουμε την επαλήθευση. Πέρας. Απορρίφθηκε. Δύο Οι 160 και 161, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεν είναι σαφέ ούτε και αυτό το αποτέλεσμα. Αυτές οι δύο παρακαλώ οι τροπολογίε να τι ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρασα. Εγκρίθηκαν. Σύμβαστε και 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Να ψηφίσουμε παρακαλώ και ηλεκτρονικά για να επαληθεύσουμε την 176. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 191. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Επαλήθευση για την 13, ε, παρακαλώ. Έναρξη. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκριθηκε. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά 17, 22 λοιπόν υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται 23 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται 24 23 παρακαλώ να την επαληθεύσουμε. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται και είχατε δίκιο. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Πάμε κατευθείαν στην 27, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 27, αν και νομίζω ότι απορρίφθηκε. Αλλά θα ελέγξουμε. Πέρας. Μα ναι, φυσικά και απορρίπτεται, αλλά δεν σηκώνετε τα χέρια σα. Συμβαστική 4, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Έγκρινεται. Συμβαστική 6, υπέρ. Κατά. Άποχε. Έγκρινεται. Και τώρα να περάσουμε κατευθείαν στην τελική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας.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 Le rapport de Madame Ayuto. Έκθεση Αγιούτου, λέει ο Πρόεδρος. Εντάξει, κύριε Αγιούτου. Allez, nous commençons. Compromis 1. Συμβαστική, υπαριθμόν 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Compromis 2, qui est pour. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές,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 Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα κάνουμε επαλήθευση. 28. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 154. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32-33. Συγγνώμη, διορθώνει πρόεδρος, 31-32. Το έκανα επίτηδες να δω εάν παρακολουθείτε. Ψηφίζουμε υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές και ψηφίζουμε. Την 31 και την 32. Ένας παραπάνω από τους σοσιαλιστές. Επαλήθευση και απορρίπτεται. 13. Συμβαστική. Περ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική, συγγνώμη, η τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14. Συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ.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 Κύριε Φαντεκάμπ, ε, έχετε το ίδιο κείμενο μπροστά σας όπως εγώ. Ωραία. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την συμβαστική 21. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ Α, όχι, συγγνώμη, το 53 καταπίπτει και πάμε στο 58. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ κατά αποχές. Νομίζω απορρίπτεται επαλήθευση. Δεν πειράζει, δεν πειράζει κύριε Ντυρό. Δεν πειράζει. Τη δουλειά γίνεται από τη συσκευή. Πέρα ψηφοφορία. devoir. 66. Qui est Πάμε στο 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Για το 66. Ψηφίζουμε πέρας. Απορρίπτεται. Όπως σας είπα. Δεν με πιστεύετε. 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 67 ε, υπέρ κατά 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται επαλήθευση ψηφίζουμε για το 69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 Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Συγχαρητήρια κυρία Αγιούτο, με ευρία πλειοψηφία εγκρίνεται το κείμενό σας. Και τώρα πάμε στην εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Ψηφίζουμε την εντολή προς διαπραγματεύσεις. Ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται. Ετοιμαστείτε για διαπραγματεύσεις, κυρία Αγιούτο. Et nous continuons. Παρακάτω. Avec. Donc, Madame Ayuto, Et là, on est sur... Monsieur Et nous continuons avec le rapport de... Συνεχίζουμε με την έκθεση ΡΙΚΕ. Έτοιμοι. Πάμε. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. ECR. Κάνετε πολύ φασαρία. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38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 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 45 όχι έχει αποσυρθεί όπως και το 10 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στο 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επαλήθευση για το 58 Le vote est clos. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, απασχόληση, Επιτροπή Απασχόλησης 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επιτροπή Απασχόλησης 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται για την ε, συμβαστική 3 επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Ah bah, il lève pas la main, hein. Tu te rends compte là Allez, on continue. Παρακάτω. Δύο ταυτόσημες. 66-67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν καταλαβαίνω τι ψηφίζετε γιατί δεν σηκώνετε το χέρι. Κύριε Φαντεκάμπ, βρισκόμαστε στις ταυτόσημες 66-67. Ταυτόσημες, είστε έτοιμος. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Ψηφίζουμε πέρας. Εγκρίνονται. 4. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απασχόληση. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το 15. Allez, je vais fermer le vote. Le vote est clos. Πέρα Εγκρίνεται. Πέντε υπέρ. Συγγνώμη, συμβαστική πέντε διορθώνει πρόεδρος, υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 19, υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 20, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 21, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2, ταυτόσημες, 22 και 23, υπέρ, αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα και επαλήθευση για αυτές τις δύο τις τρεις γιατί έχουμε μαζί και την έμπλ 1 προσθέτει πρόεδρος πέρας ψηφοφορίας εγκρίνονται 24 υπέρ κατά αποχές Έγκρινονται. 26 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 25 καταπίπτει έμπλ 2 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ θέλετε επαλήθευση για την έμπλ 2 ψηφίζουμε ψηφίζουμε Πέρας. Εγκρίνεται. 6. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, λόγη παράγραφος 10 β νέο. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Ψηφίζουμε. Πέρας. Πήρετε 40 ψήφου υπέρ και συγχαρητήρια με ευρία πλειοψηφία εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για την εντολή προ διαπραγματεύσει. Ψηφίζουμε. Πέρα. Εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία η εντολή. Συγχαρητήρια κύριε Ρικέ. Άλλη μια έκθεση λοιπόν. Δύο μάλλον εκθέσει του Πίπερ για τον ανταγωνισμό στον, στις αερομεταφορές. Πρόκειται για ψηφοφορία ε, Τελική ψηφοφορία λοιπόν για την έκθεση του κυρίου Πίπερ. Πέρασε. Συγχαρητήρια στην κύριο Πίπερ. Με μεγάλη πλειοψηφία κρίνει. Το ίδιο λοιπόν ψηφοφορία επαλήθευση της έκθεσης της κυρίας Μάισνερ για τα αποβλητά των πλοίων. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρας. 46 η ψήφη υπέρ, καμία αποχή, καμία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια στην κυρία Μάισνερ και για όσους θα μας αφήσουν να πω ότι ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίε και έτσι θα περάσουμε στην Σύμβαση για την Επιτροπή για την Κοινότητα Μεταφοράς. Αν θέλετε παρακαλώ να εξέλθετε τις αιθούσεις ήσυχα. Θέλετε διάλειμμα. Ένα λεπτό διάλειμμα παρακαλώ. Nous reprenons nos travaux, s'il vous plaît. Et nous sommes... επανέλθουμε στις εργασίες, στις εργασίες μας και είμαστε στο υπαριθμό 19, θέμα της ημερησίας διατάξεως. Έχουμε βεβαίω πάλι σύντα την κυρία Ντελή, δηλαδή εμένα προσωπικά. Ε, στην έκθεση αυτή περί τίνος πρόκειται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 είχε προτείνει διαπραγμάτευση συμφωνίας για ρυθμίσεις, για ε, τεχνικά πρότυπα που θα εφαρμόζονταν από τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων που να είναι συμβατά με τις ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Και στην βάση της θετικής εμπειρίας από την εφαρμογή των συνθήκων της κοινότητας ενέργειας για τη δημιουργία κοινότητας μεταφορών, οδικών, σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών οδών και θαλασσίων και δικτύων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Δυτικών Βαλκανίων. Συμφωνία για τη δημιουργία κοινότητας μεταφορών με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα έχουν επιπτώσει στην καθημερινή ζωή των πολιτών και ιδίως ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια ή για παράδειγμα ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια. Με την εγγύηση μεγαλύτερης ασφάλειας και προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή αυτή, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη. Η ε, συνθήκη αυτή θα βοηθήσει τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων να ευθυγραμμίσουν τι σχετικέ νομοθεσίε του με αυτές τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Κάτι το οποίο θα ενισχύσει τι ε, σχέσεις γειτονίας, τις διαμεθοριακές συνεργασίες και θα φέρει πιο κοντά τις χώρες αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η συνθήκη αυτή που ιδρύει η κοινότητα μεταφορών υπεγράφει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2007 υπό την επιφύλαξη ολοκλήρωσης σε απότερο χρονικό διάστημα με όλη τη συμμετοχή όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων εκτός του Κωσόβου που έχουν ήδη κυρώσει την συνθήκη η οποία εφαρμόστηκε προσωρινά μεταξύ των μερών. Εν ώψη των ε, γεγονότων αυτών προτείνουμε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού να τοποθετηθεί θετικά για την ολοκλήρωση της συνθήκης αυτής. Ανοίγουμε τώρα τον διάλογο με τους σκιώδεις εισηγητές. Κύριε Ντέλη, καλημέρα σας. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, δεν έχω πολλά να πω, λέει ο κύριος ε, Ντέλη. Θεωρώ ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων χρειάζονται περισσότερο συντονισμό στον τομέα των μεταφορών, στρατηγικών υποδομών, θέσπισης προτεραιοτήτων. Είναι γνωστό ότι σημειώνονται σημαντικέ εντάσει μεταξύ των χωρών τη περιοχής αυτής και τώρα ακόμη μετά από τόσα χρόνια, αλλά είναι και μια περιοχή όπου οι πρωτεύουσε των χωρών αυτών δεν διασυνδέονται ούτε με αυτοκινητοδρόμους, ούτε με σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει και πρέπει να βελτιωθεί η περιφερειακή συνεργασία. Και για να γίνει αυτό πρέπει να προωθήσουμε τις υποδομές μεταφορών και όλα τα άλλα δίκτυα επικοινωνιών, αλλά και προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή αυτή. Άρα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει απολύτως την έκθεση. Σας ευχαριστώ και εντελή, λέει η κυρία Ντελή. Ε, κυρία Ντεμόντε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα, μπράβο για ε, τα όσα έγιναν και συμφωνώ ε, ότι είναι σημαντική αυτή η περιοχή. Πρόκειται περί χώρες που είναι κοντινές και επίκειται η ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική συγκυριακή είναι παγίως ε, μπερδεμένη και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με υποδομές σε σχέση με τις μεταφορές. Αυτό αποφασίστηκε το 2015 να επεκταθούν δηλαδή τα TNT και θα πρέπει επομένω όλα αυτά να λάβουμε υπόψη. Πρόκειται για τον διάδρομο Ανατολικής Μεσογείου. Θα πρέπει Ευρωπαϊκή Ένωση να προσέξει το πώς θα αναπτυχθεί η υπόθεση των υποδομών εκεί στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό από την Κίνα. Είναι η κατάσταση λεπτή, έχουν αναπτυχθεί διπλωματικές δραστηριότητες και άρα επομένω το Βερολίνο ήταν μια επιτυχία Επίσης ε, και στις 12 Ιουλίου του 2017 συνάντησε κορυφής της ε, ταιριές της όπου και υπεγράφει εν λόγω συμφωνία και ε, αποφασίστηκε να καλυφθεί η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Γιατί υπήρχε πρόβλημα σχετικά με την Προεδρία, υπήρχαν κάποιες περιπλοκές όσον αφορά τους σειροδρόμους. Πάντως, πάντως, προσυπέγραψαν την ε, συμφωνία και οι Βόσνοι και έτσι ε, καθίσταται ευκολότερη η προσέγγιση. Υπάρχουν ακόμα κάποια καθόδη ζητήματα, το κοσυφοπαίδιο, ε, προστρεβή με την Σερβία. Ε, πάνω το δούμε αισιόδοξα, εν μέρη έχει ξεπεραστεί και το πρόβλημα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας επίσης και πρόκειται επομένως για σημαντική συμφωνία και όπως επανειλημμένα είπε η Πρόεδρος χρειάζεται να εμπλακεί πιο δραστήρια, πιο ενεργά το Κοινοβούλιο. Πρόκειται για διακυβερνητική λειτουργία. Όμως ε, θα πρέπει ε, κατόπιν της ε, συνήξης της Λισαβόνας να δικαιούται να εμπλακεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε, οπωσδήποτε, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για συναντήσεις όπως έγινε και πριν από δύο χρόνια στην Πριστίνα. Και έτσι το Κοινοβούλιο να δει τι ισχύει επιτόπου από πλευράς πολιτικής, από πλευράς ε, υποδομών, γιατί πρόκειται για χώρες που είναι στα πρόθυρα της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, να βοηθήσουμε, να έχουμε διαγενοβουλευτικές ε, επαφές, συνεργασία και με την ΑΦΕΤ. Οι δύο επιτροπές μας είναι πολύ σημαντικές όσον αφορά την πρόοδο της υπόθεσης. Μεταφορές και υποδομές είναι σημαντικές μεταβλητές για την εξωτερική πολιτική. Άρα θα πρέπει αυτό το κείμενο να εγκριθεί και τώρα κατά τα τέλη της θητείας να αναδείξουμε το πόσο σημαντική είναι μια τέτοια προσέγγιση και με τη νέα θητεία να έχουμε ακόμα πιο αποφασιστική ε, ε, αντιμετώπιση πολιτική και ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο. Κύριε έχει το λόγο. Πρόεδρε, δεν είμαι σκιώδης εισηγητής από το ECR, αλλά το θέμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε πάρα πολύ στο τεκτενόμενα στην περιοχή αυτή, γιατί η περιοχή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και τη δική μας ομάδα και θεωρώ ότι και η ομάδα μας θα μπορέσει να υποστηρίξει απόλυτα την ε, έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μάκερ. Θα πρέπει να εξετάσετε το θέμα αυτό με την γραμματεία, γιατί εγώ σας έχω καταχωρισμένο ως σκιώδης, γιατί αν δεν είστε εσείς ο σκιώδης, πείτε μου ποιος είναι σκιώδης από την ομάδα σας. Ευχαριστώ. Να το κοιτάξω, πρόεδρε, θα το κοιτάξω. Ο κύριος Τελίνσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδη. Ο κύριος Ράντος όμως δεν μπορεί να παραπευθεί σήμερα. Μου ζήτησε λοιπόν να πάρω το λόγο εξ ονοματό του. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι σαφής γιατί ήδη μίλησα σήμερα, ζητήσα ε, ένα μικρό διάλειμμα και εσείς το ερμηνεύσατε ως ε, αίτημα αναβολής ε, της ψηφοφορίας. Να μιλήσω αργά για να με καταλάβετε. Εξ ονοματός του κύριου Ράντος. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τον εισηγητή που μας παρουσίασε το σχέδιο ε, πρόταση σε ό,τι αφορά την πρόταση του Συμβουλίου. Θα ήθελα, ο συνάδελφος να τονίσει ότι η σύμβαση αυτή έχει ως σκοπό να ε, βοηθήσει τις μεταφορές μεταξύ των Δυτικών Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενδυναμωθεί και η διαδικασία προσχώρησης των Δυτικών Βαλκανίων και έτσι έχουν ήδη προκύψει θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία και η, επέκταση λοιπόν του ΤΕΝΤΗ στην Βυτική, στα δυτικά Βαλκάνια το 2016, η ατζέντα της συνδεσιμότητας ανοίχθη σε μια κορυφαία προτεραιότητα για τη χώρα. Έτσι διευκολύνεται η επαφή μεταξύ των ε, ανθρώπων και η επανασυμφωλίωση σε ό,τι αφορά και την προοδευτική ενσωματώση των αγόρων και την ένταξή του ε, στην ε, Ευρώπη. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι υποστηρίζουμε πλήρως μαζί με τον κύριο Ράντο στην θέση του εισηγητή ότι η Επιτροπή Τραν θα πρέπει να δώσει θετική γνώμη για την σύναψη τη συμφωνίας της σύμβασης και να κάνετε και κάποια σχόλια εξ ονόματός μου ω συντονιστή μιας και μία φράση στις δύο εβδομάδε είμαι στα Δυτικά Βαλκάνια. Ποια είναι η προσωπική μου εντύπωση για την ε, υποδομή. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πλεονέκτημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κινηθούμε προ την κατεύθυνση αυτή. Πρόκειται για μια κατάσταση που θα πρέπει να βελτιωθεί και χαίρομαι που θα υπάρξει διόρθωση με τον τρόπο αυτό. Σα υποστηρίζω λοιπόν, Πρόεδρε, και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τρίτσκα. Αν δεν θέλει κανείς άλλο να πάρει το λόγο. Να στραφώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δώσω το λόγο στον κύριο Μπαρόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστηρίζω και τονίζω την εκτίμησή σας, κυρία Πρόεδρε, και αυτές των σκιωδών σε ό,τι αφορά τη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής. Όπως όλοι σας είπατε, πολύ εύστοχα. Το θέμα τη συνδεσιμότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, ευημερία. Και τα Δυτικά Βαλκάνια περιτριγυρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα είναι λογικό να εισαχθούν στην έννοια αυτή Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό και στις ε, μεταφορές. Η Επιτροπή Μεταφορών λοιπόν θέλει να δημιουργήσει μια νέα ορμή σε ό,τι αφορά τα Βαλκάνια, γιατί η κοινότητα μεταφορών ενδυναμώνει τους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προβολιάνοντας το έδαφος για τη μελλοντική προσχώρηση. Με τους συναδέλφους μας λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι για την ε, κοινότητα μεταφορών και η επιτυχία αυτής ε, εξαρτάται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι μεταφορέ που βρίσκονται στο επίκεντρο τη ζωή και των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων μπορεί να μα βοηθήσουν να πετύχουμε αυτή τη συμφωνία. Η κοινότητα μεταφορών ε, συνοδεύεται και από τη στρατηγική για τα Βυτικά Βαλκάνια που ορίστηκε στι αρχέ του 2018 για να δημιουργηθεί μια νέα υποστήριξη και νέα κίνητρα για την περιφέρεια. Θέλουμε λοιπόν πλήρη εφαρμογή τη ε, κοινότητας μεταφορών και των ε, εντοπισμένων στόχων πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε βεβαίως την πρόταση της Επιτροπής σας και από εσάς προσωπικά κυρία Πρόεδρε και την υποστήριξη που εκφράζεται για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια σας. Πρόθεσμια για τα τροπολογιών. Σας υπενθυμίνω. Είναι η 16η Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι. Και να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για μια διαδικασία έγκρισης Και άλλα Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση. Σε 5 έω 8 λεπτά θα ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ένα μικρό λοιπόν διάλειμμα για να καταφτάσουν οι συντονιστές. Και έτσι λοιπόν έχουμε ένα μικρό διάλειμμα για 8 λεπτά. Nous devons être revenus 12 και 3 παρακαλώ.